Vi prego di prendere posto. Παρακαλώ να καθίσετε. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε με τις ψηφοφορίες. Ha chiesto la parola onorevole Marias. O κύριος Μαριάς. Per un punto all'ordine del giorno. La parola onorevole Marias. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, στις 17 Δεκεμβρίου το Κοινοβούλιο μας έκανε δεκτό ψήφισμα με το οποίο καταδίκαζε τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπουρούντι και ζητούσε την άμεση απελευθέρωση του Έλληνα υπηκόου Σπύρου Ρίτσαρτ Χαγκαμπιμάνα, ο οποίος είχε φυλακιστεί στα τέλη Ιουνίου, γιατί σαν επικεφαλής αστυνομικός αρνήθηκε να δώσει εντολή στις δυνάμεις καταστολής να πυροβολήσουν κατά των διαδηλωτών. Θέλω να ενημερώσω λοιπόν σήμερα το σώμα για το αίσιο τέλος της περιπέτειας του Σπύρου, ο οποίος την προηγούμενη Παρασκευή 15 Ιανουαρίου κρίθηκε αθώος από το δικαστήριο και σύντομα θα είναι ελεύθερος για να βρεθεί κοντά μας. Η εξέλιξη αυτή αποδεικνύει τη σημαντική επιρροή που μπορεί να έχουν οι αποφάσεις του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να συνεχίσουμε αταλάντευτοι. ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Μαριά. Είμαι πεπισμένος ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε και θα συνεχίσει να έχει σημαντικό ρόλο και βάρος μιας και εκπροσωπεί 550 εκατομμύρια ε, ψηφοφόρους, πολίτες μάλλον. Ας ξεκινήσουμε με την έκθεση Χάουταλα, άρση ασυλίας του Τσέσλα Φάνταμ Σεκίρσκι. είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. η δεύτερη έκθεση Χάουταλα, η δεύτερη αίτηση άρση ασυλίας του κυρίου Σεκεύσκη. Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά, αποχές, δεκτή. Συνεχίζουμε τώρα με την έκθεση ΜΑΤΟ για το πολιετές σχέδιο αποκατάστασης του Ευηθοπτέριου τόνου στην Ανατολική Μεσόγειο ψηφοφορίες 1 με 40 ομαδών. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτές. Άρθρο 8. Μετά την παράγραφο 6 τροπολογία 41. Ονομαστική ψηφοφορία ψηφίζεται. La votazione è chiusa. Πέρα της ψηφοφορίας. Δεκτό. Μετά από πρόταση τώρα της, ε, την πρόταση της Επιτροπής περ κατά, αποχές, δεκτή. Θέλει το λόγο εισηγητής. Κύριε Μάτο, έχετε ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα μόνο να ζητήσω από το Κοινοβούλιο να μην εγκρίνει το μαθητικό ψήφισμα για να αρχίσουν αμέσως οι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν τώρα μετά από την πρόταση του εισηγητή ζητά να μην ψηφιστεί η πρόταση νομοθετική. Ποιοι είναι υπέρ της πρότασης του εισηγητή, ποιοι είναι κατά, ποιοι απέχουν. Συνεπώς γίνεται δεκτή η πρόταση ΜΑΤΟ. Το θέμα λοιπόν παραπέμπεται στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Περνάμε τώρα στην έκθεση Λάγκεν, ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. ή 7. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. <coughs> Απορρίπτεται. Παράγραφος 5. Αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για το δεύτερο τμήμα. La votazione è chiusa. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 9 το αρχικό κείμενο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για το 9. Ψηφίζεται. Πέρα στις ψηφοφορίες. Απερίφθη. Παράγραφος 14. Αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές δεκτό τροπολογία 11 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή 13 υπέρ κατά Αποχές. Απορρίπτεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 21 αρχικό κείμενο υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. 35 αρχικό τμήμα το πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές δεκτό ηλεκτρονικός έλεγχος για το δεύτερο τμήμα του τμήματος 35 ψηφίζεται La votazione chiusa. Πέρα στις ψηφοφορίες. Παράγραφο 41 αρχικό κείμενο υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. 46 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. 54 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. Μετά την 54 έχω την 15, τροπολογία 15 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη αρχικό κείμενο 60 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. 61 αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. 63 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές δεκτό δεύτερο τμήμα υπέρ άρχεται μάλλον ε, η ψηφοφορία ηλεκτρονική ψηφοφορία τέλος δεκτό το κείμενο της 63 65 αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές 18 66 αρχικό κείμενο σε τρία τμήματα πρώτο υπέρ κατά αποχές δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές δεκτό. Τρίτο τμήμα υπέρ, α, θα υπάρξει ηλεκτρονικός έλεγχος για το δεύτερο τμήμα του 66. Τέλος. Απερίφθη. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές δεκτό 73 σε δύο τμήματα πρώτο υπέρ κατά αποχές δεκτό δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό 75 υπέρ κατά αποχές Ηλεκτρονικός έλεγχος για το αρχικό 75. Ψηφίζεται. Πέρα στις ψηφοφορίες. Απερίφθη. 76 σε τρία τμήματα. Πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές δεκτό. Τρίτο τμήμα ονομαστική ψηφοφορία ψηφίζεται. Πέραση ψηφοφορίας. Δεκτό. 78 αρχικό υπέρ κατά αποχές δεκτό. 81 αρχικό σε δύο τμήματα πρώτο υπέρ κατά αποχές δεκτό δεύτερο τμήμα ονομαστική ψηφίζεται Πέραση της ψηφοφορίας δεκτή 84 σε τρία τμήματα πρώτο υπέρ κατά αποχές δεκτό δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό τρίτο τμήμα υπέρ κατά Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για το τρίτο τμήμα. Ψηφίζεται. Πέρα τη ψηφοφορία το κείμενο γίνεται δεκτό. 86 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Ηλεκτρονικός έλεγχος ξανά για το 86 ψηφίζεται. Τέλος της ψηφοφορίας. Απερίφθη. Παρακαλώ να σηκώνετε τα χέρια γιατί δεν μπορώ να δω. 87 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος και για το 87. Πέρα της ψηφοφορίας το 87 γίνεται δεκτό. 88 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. 89 υπέρ, ονομαστική ψηφοφορία μάλλον. Για το 89 ψηφίζεται. Τέλος της ψηφοφορίας. Δεκτό. Μετά την παράγραφο 89 έχω την τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Παράγραφος 94 υπέρ κατά αποχές δεκτό. Μετά την 99 έχω την τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές δεκτό. Παράγραφος 104 υπέρ κατά αποχές δεκτό. 105 αρχικό υπέρ κατά αποχές δεκτό. 106 αρχικό υπέρ Ηλεκτρονικός έλεγχος ζητήθηκε για το 105. Ψηφίζεται. Πέραση ψηφοφορίας. Δεκτό. 106 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για το 106. Νομίζω ότι έχει απορριφθεί αλλά ας το ελέγξουμε. Ψηφίζεται. Τέλος της ψηφοφορίας. 107 αρχικό υπέρ κατά αποχές δεκτό 111 υπέρ κατά αποχές δεκτό 112 υπέρ κατά αποχές δεκτό 113 υπέρ κατά αποχές δεκτό Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 4 ητά αποχές δεκτή. Λοιπόν με το H αγγλικό υπέρ κατά αποχές δεκτό. P αγγλικό υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για το P αγγλικό. Τέλος, δεκτό το π. Μετά έχω το Q, την τροπολογία 5. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για το, την τροπολογία 5 παρακαλώ. Τέλος. Απερίφθη. 6. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Σύνολο του ψηφίσματος τροπολογημένο. Ονομαστική ψηφοφορία ψηφίζεται. Τέλος της ψηφοφορίας. Συγχαρητήρια κύριε Λάγκεν. Περνάμε τώρα στην έκθεση World. Διαπολιτισμικός διάλογος. Υπάρχει μια πρόταση ψηφίσματος εναλλακτική, είναι η τροπολογία 1. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. Παράγραφος 7 τώρα, το αρχικό κείμενο. Κοιτάξτε, ήταν σαφής η πλειοψηφία, λέει ο Πρόεδρος, αλλά αν θέλετε, αν επιμένετε, ας υπάρξει έλεγχος για την 1. Ψηφίζεται. Πέρα στις ψηφοφορίες δεν υπήρξαν σχόλια από ό,τι ακούω. Παράγραφος 7. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές δεκτό δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ηλεκτρονικός έλεγχος για το δεύτερο τμήμα τέλος της ψηφοφορίας απερίφθη Λοιπόν, συνολικά το απολογημένη, ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζεται. Τέλος. Το κείμενο γίνεται δεκτό. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Έχεις δει στο λόγο. Συγήτρια, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους τους συναδέλφους, λέει κύριε Γουόρτ, και ε, όλα ε, τα μέλη του προσωπικού, εμπειρογνώμονες για τα θέματα του πολιτισμού, ομάδες θρησκευτικέ, τους νέους, όλους όσοι με βοήθησαν να συντάξω μια έκθεση που δίνει μια θετική εικόνα για το μέλλον, για τους νέους, για τις μελλοντικές κοινότητες σε μια διαδικασία ε, διαλόγου και συνεννόησης. Αυτό είναι ο διάλογος. Συζητήσεις, συνεννοήσεις. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, περνάμε τώρα στην έκθεση παλτς ε, σχετικά με τις ε, προκλήσεις που έχουν σχέση με τα χρηματοπιστωτικά θέματα. Παράγραφος 2. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αρχικό κείμενο η 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 24 σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 26 σε δύο τμήματα αρχικό κείμενο, πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 26 αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 59 αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά απο... εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ε, εδάφιο α σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, επίσης πάμε τώρα στην ονομαστική ψηφοφορία για το σύνολο του ψηφίσματος υπέρ παρακαλώ. Ηλεκτρονική ψηφοφορία έκλεισε. Εγκρίνεται το κείμενο. Συγχαρητήρια στον συνάδελφο κύριο Μπάλτ. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα ε, στις ε, ε, Γενική επιχειρηματικότητα παράγραφος 1 αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η πέντε αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται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 αποχές εγκρίνεται. Η 22 αρχικό κείμενο ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίθηκε το κείμενο, η 29 αρχικό κείμενο υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 30 αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 36 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, αιτιολογική σκέψη G, D, μάλλον υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, ε, αιτιολογική σκέψη το αρχικό κείμενο G, πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, το L ε, πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το X λατινικό αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη Z λατινικό αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα με ονομαστική ψηφοφορία για το σύνολο του κειμένου του ψηφίσματος. Ε, ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται το κείμενο. Συγχαρητήρια στη συνάδελφο κυρία Ματέρα. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Έκθεση πλούρα πολιτικές δεξιοτήτων για την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας.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 αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η εννέα, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η δεκατέσσερα, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η δεκαεπτά, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Λοιπόν, ηλεκτρονική επαλήθευση για την 20. Έκλεισε η ψηφοφορία, απορρίφθηκε το κείμενο. 21 σε τρία τμήματα. Πρώτο, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ή το δεύτερο, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τρίτο, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 22, δύο τμήματα. Πρώτο, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 24, δύο τμήματα. Πρώτο, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 33, δύο τμήματα. Πρώτο, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 34. Δύο τμήματα. Πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 49 σε δύο τμήματα πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 50, δύο τμήματα, πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, δεύτερο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 51, δύο τμήματα, πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, δεύτερο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 54, υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται η 60 δύο τμήματα πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 62 αρχικό κείμενο πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ή 6 μισό λεπτό ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. 63. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Ε, κοιτάξτε, είχα την εντύπωση ότι επαληθεύσαμε το δεύτερο του 63 γιατί στην οθόνη δεν ξέρω, άλλα έδειχνε. Ε, τι ψηφίσαμε λέει ο πρόεδρος, ε, ψηφίσαμε τώρα, θέλετε να επαναλάβουμε. Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε. Ήταν σαφές, ψηφίζαμε για το δεύτερο τμήμα. Αυτό είχατε ζητήσει. Ψηφίζουμε τώρα, ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίζουμε για το 62 δεύτερο τμήμα. Παρακαλώ. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίθηκε το κείμενο. Η 63 Αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 64. Υπέρ κατά αποδίνεται. 65. Υπέρ κατά αποχές 63. 66. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 67. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 68. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 69 δύο τμήματα πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 72 τμήματα πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ε, το G, αιτιολογική σκέψη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το M, δύο τμήματα, πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, δεύτερο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Q, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. R, λατινικό, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. S, λατινικό, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Λοιπόν, τώρα ψηφίζουμε για το σύνολο του ψηφίσματος, μονομαστική ψηφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. La votazione chiusa. Έκλεισε η ψηφοφορία. Τώρα, το κείμενο εγκρίθηκε. Συγχαρητήρια στον εισηγητή κύριο Πλούρα. Και περνάμε στην έκθεση την τελευταία Κάλλας Γκίπχαρτ που είναι ε, προς μια νομοθετική πράξη για την ψηφιακή ενιαία αγορά. 1.14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 5 υπέρ κατά αποχές απερίφη. 24 υπέρ κατά αποχές απερίφη. Αρχικό κείμενο 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 1. Πέρα της ψηφοφορίας. Απερίφθη. Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 15 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 16 υπέρ σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Δεκτό, λάθος λέει ο πρόεδρος. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για το δεύτερο της παραγράφου 16 Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. Δεκτό. 19 αρχικό υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 30 σε 3 τμήματα πρώτο. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές δεκτό. Τρίτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές δεκτό. 31 δύο τμήματα πρώτο υπέρ, κατά, αποχές δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές δεκτό. 34 σε δύο τμήματα πρώτο υπέρ, κατά, αποχές δεκτό. Δεύτερο τμήμα ονομαστική ψηφοφορία, δεύτερο του 31. Πέρας της ψηφοφορίας. Δεκτό. 35 σε δύο τμήματα υπέρ. Πρώτο, κατά, δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονικός έλεγχος. Για το δεύτερο τμήμα της 35. Τέλος της ψηφοφορίας δεκτό. 21 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 22 υπέρ αποχές απερίφθη. 47 σε 2 τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτή. Δεύτερο τμήμα ονομαστική ψηφοφορία. Δεύτερο τμήμα 47. Τέλος ψηφοφορίας δεκτό. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Καταπίπτει το αρχικό 53. Θέλετε να υπάρξει ηλεκτρονικός έλεγχος για την παράγραφο 53 ή για την 25. Για την 25 ηλεκτρονικός έλεγχος. Την τροπολογία εννοείται 25 ηλεκτρονικός έλεγχος. Πέρα στις ψηφοφορίες. Δεκτό. Καταπίπτει λοιπόν το παλαιό 53. Περνάμε τώρα στην 56 τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Αρχικό 59 σε δύο τμήματα. Πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Δεύτερο τμήμα ονομαστική ψηφοφορία. Τέλος. Δεκτό. 62 σε δύο τμήματα. Πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Δεύτερο τμήμα ονομαστική. Τέλος. Δεκτό. 63. Αρχικό κείμενο στο πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό. 64 σε δύο τμήματα. Το πρώτο ονομαστική ψηφοφορία για το πρώτο τμήμα της παραγράφου 64 ψηφίζεται. Τέλος. Δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 23 ονομαστική ψηφοφορία. Τέλος. Απερίφθη. Λοιπόν, ονομαστική ψηφοφορία για το 65, ποιοι είναι υπέρ, μάλλον ονομαστική ψηφοφορία, τέλος της ψηφοφορίας δεκτό. 67 ονομαστική ψηφοφορία ψηφίζεται. Τέλος. Δεκτό. 68. Ονομαστική ψηφοφορία ψηφίζεται. Εβδομήντα Αρχικό σε δύο τμήματα. Πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. 73 αρχικό σε δύο τμήματα πρώτο υπέρ κατά αποχές δεκτό υπέρ κατά αποχές δεκτό και το δεύτερο τροπολογία προφορική μπερές στην 76 Α, όχι δεν υπάρχει. Οπότε ψηφίζουμε την τροπολογία 26. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή.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 κατά, αποχές, δεκτό. Τροπολογία 2 τώρα, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. 89 θέλετε να γίνει ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 2. Ψηφίζουμε λοιπόν ηλεκτρονικά για την 2. Μετά την παράγραφο 88.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 Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. Μετά την παράγραφο 100 υπάρχει η τροπολογία 7 υπέρ, κατά, αποχές, δε, Τροπολογία 8 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. Ε, παράγραφος αρχική 110 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Τροπολογία 17 υπέρ, κατά,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 10 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Τροπολογίες 3 και 11 στην 125. Έχει ζητήσει το λόγο η συγγήτρια. Ναι. Μου επέστησαν την προσοχή ότι σε αυτή την τροπολογία η γαλλική μετάφραση είναι λάθος και λέει ακριβώς το αντίθετο από το αρχικό κείμενο που είναι το αγγλικό. Το αγγλικό κείμενο ψηφίζουμε και όχι τη λάθος γαλλική μετάφραση παρακαλώ. Ήθελα μόνο να σε επιστήσω την προσοχή σε αυτό. Θα δούμε αν έχουν υπάρξει λάθη και θα τα διορθώσουμε. Ψηφίζουμε τώρα τις τροπολογίες 3 και 11 στο αρχικό κείμενο. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτές. 19 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. 20 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη απερίφθη 12 θέλετε να υπάρξει για την τροπολογία 20 ε, ηλεκτρονικός έλεγχος ψηφίζετε λοιπόν για την 20 ηλεκτρονικά τέλος 72 υπέρ 130 κατά Κοιτάξτε, με βάζετε να ψηφίζω ενώ είναι ξεκάθαρο το αποτέλεσμα και χάνουμε χρόνο όλοι. Λοιπόν, τροπολογία 12. Υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. 13 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. Ψηφίζουμε τώρα το ψήφισμα στο σύνολό του ονομαστική ψηφοφορία. La Πέρα τη ψηφοφορία, συγχαρητήρια, δεκτό το κείμενο, κάνατε πολύ καλή δουλειά. Περνάμε τώρα στις επεξηγήσεις ψήφου.